Αξιότιμη Γενική Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, είναι μεγάλη μας χαρά να σας καλωσορίσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκ νέου. Αξιότιμη κυρία Μπαν, και προς εσάς, ε, σας, ε, κυρία Μπαν, σας καλωσορίζουμε και εσά εδώ που συνοδεύσατε τον ε, σε δικό σας σήμερα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Σας καλωσορίζουμε. Πριν από 70 χρόνια, κυρία Γενικά, Γενική Γραμματέα, το 1945, στο Σαν Φρανσίσκο ιδρύθηκαν τα Ηνωμένα Έθνη. Σήμερα, αξιότιμε κύριε και κύριοι, τα Ηνωμένα Έθνη είναι η πιο σημαντική οργάνωση της διεθνούς συνεργασίας. Πρόκειται για τον πυλώνα, τον φέροντα πυλώνα της παγκόσμιας και μια οργάνωση απαραίτητη για τη διατήρηση της διεθνούς ασφάλειας. Και για την διεθνή ασφάλεια αυτή υπάρχουν πολλές προκλήσεις παντού στον κόσμο, όπως ποτέ πριν, ποτέ άλλοτε. Και γι' αυτό τον σκοπό λοιπόν τα Ηνωμένα Έθνη διατραματίζουν σημαντικό και κεντρικό ρόλο για την επίλυση των συγκρόσεων και πρέπει να πρόκειται για ένα απαραίτητο εργαλείο για την εξέβρεση ειρηνικών λύσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα το Κοινοβούλιο αυτό συμμερίζεται τους στόχους της οργανωσής σας, κυρία Γενική Γραμματέα, την καταπολέμηση των συνέπειων της αλλαγής του κλίματος, η καταπολέμηση κατά της φτώχειας και της πείνας, η δέσμευση για την εκπαίδευση και τη βιώσιμη ανάπτυξη, μόνο αυτή οι στόχοι αποτελούν τους βασικούς, τις βασικές προϋποθέσεις για τις ειρηνευτικές διαδικασίες. Για τις ειρηνευτικές διαδικασίες, τις οποίες όπως ανέφερα χρειαζόμαστε κατεπηγόντως εδώ λοιπόν ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορώ χωρίς ε, επιφύλαξη να σα πω εξ ονόματο όλων των συναδέλφων ότι σα υποστηρίζουμε και γι' αυτό λοιπόν είναι μεγάλη τιμή που σα ε, καλώς ορίζουμε εδώ στον οίκο τη Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είναι η δεύτερη φορά που σας καλωσορίζουμε και σας δίνουμε το λόγο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σα παρακαλώ, έχετε το λόγο. Your κύριε Πρόεδρε Σούλτς, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριοι Επίτροποι, κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που μπορώ να απευθύνω το λόγο στους αντιπροσώπους των ευρωπαϊκών λαών. Συγχαίρω καταρχάς τον πρόεδρο Σούλτς, στον οποίο αποδεμήθηκε το βραβείο Καρλομάγνου πριν λίγες μέρες, για το ρόλο του στα πλαίσια της προώθησης της δημοκρασίας στην Ευρώπη και γιατί έφερε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιο κοντά στον Ευρωπαϊκό λαό, τον οποίο υπηρετεί. το κοινοβούλιο αυτό αντιπροσωπεύει μια μεγάλη ποικιλία πολιτισμών, παραδόσεων, με μια κοινή πεποίθηση όμως, η οποία λέγει ότι είμαστε ισχυρότεροι και είμαστε καλύτεροι όταν συνεργαζόμεθα. Παίζεται ένα σημαντικό ρόλο και σε πολλά από τα θέματα της ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών συμμετέχετε στις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών για την ειρήνη, την ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε χωρίς την εμπλοκή, την υποστήριξη και την ενθάρρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σας είμαι θα ευγνώμονες για την αφοσίωσή σας σε αυτή την προσπάθεια. Κυρίες και κύριοι, σήμερα θα ήθελα να αναφερθώ σε τρεις συνδεδεμένες μεταξύ τους προκλήσεις και θα ήθελα την προσοχή σας σε αυτές. Πρώτον, πρόληψη του βίαιου εξτρεμισμού. Δεύτερον, αντιμετώπιση της πρόκλησης της μετανάστευσης. Και τρίτον, αηφόρος ανάπτυξη για όλο τον κόσμο. Κυρίες και κύριοι, το πρώτο θέμα οι ακραίες μορφές βίας είναι συγκεκριμένες απειλές για την ειρήνη και την ασφάλεια. Ασκείται βία εις βάρος των αμάχων από εξτρεμιστικές ακραίες ομάδες, κάτι το οποίο αμφισβητεί τις καθολικές αξίες της ειρήνης, της δημοκρατίας και της ανοχής η σκόπιμη καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι μια ύβρις για την ανθρωπότητα. Συνεπώς εγώ θα συνεχίσω να συνεργάζομαι με τα ευρωπαϊκά όργανα για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Υπάρχει ένα συνολικό πρόγραμμα δράσης των Ηνωμένων Εθνών για την αποτροπή τέτοιων μορφών βίας και θα παρουσιάσουμε την τελική μας πρόταση αργότερα ε, σε λίγους μήνες. Προσπαθούμε εμείς να προωθήσουμε σε όλες τις χώρες τον έλεγχο της διακυβέρνησης, τον σεβασμό των καθολικών αξιών και τον διάλογο ανάμεσα στις διαφορετικές κοινότητες. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ο σεβασμός του κράτους δικαίου είναι θεμελιώδες. Θα πρέπει να μην ξεχνάμε τις ειδικέ ευθύνες που έχουμε έτσι ώστε να αντιμετωπίζουμε με τέτοιο τρόπο τον εξτρεμισμό έτσι ώστε να μην χειροτερεύουμε τα πράγματα. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες επιρροής των προσωπικότητων και από τον θρησκευτικό χώρο και τον χώρο της παιδείας και του πολιτισμού. Θα πρέπει έτσι να δούμε τι απασχολεί τους νέους, ακόμα και τις νέες, να απομακρύνονται από τις απλές μορφές συμπεριφοράς και να ριζοσπαστικοποιούνται χτυπώντας τους άλλους αλλά και τον εαυτό τους πολλές φορές θυσιάζοντας και τις δικές τους ζωές. Ο βίαιος αυτός, ε, οι βίες αυτές ακραίες συμπεριφορές του Μπόκο Χαράμ, του Νταές, του Αλ Σαμπάμπ και άλλων ε, τρομοκρατικών τέτοιων ομάδων. Είναι προφανές ότι συνοδεύονται οι δράσεις αυτές από μιλίες μίσους εις βάρος κομμάτων, τμήματων της κοινωνίας, εις βάρος κοινοτήτων και μεταναστών. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να συνεργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε τις απειλές αυτές στη ρίζα τους. Αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, εδώ έρχεται το θέμα της πρόκλησης της μετανάστευσης. Είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί όλους από την Μεσόγειο στην Νότιο-Ανατολική Ασία. Χιλιάδες άνδρες, παιδιά και γυναίκες χάνουν τη ζωή τους σε παρακινδυνευμένα ταξίδια διαφυγής. Σχεδόν 1.800 ε, μετανάστες ε, πνίγηκαν στη Μεσόγειο, μια τεράστια αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο οι μισοί από αυτού οι οποίοι διασχίζουν τη Μεσόγειο φεύγουν από καταχρήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και από πολεμικές συγκρούσεις και πρέπει να τύχουν, δικαιούνται διεθνούς προστασίας ως πρόσφυγες. Η Ευρώπη πρέπει να παίξει ένα συνολικό ρόλο και θα πρέπει επίσης να αναλάβει την ευθύνη αυτή. Η διάσωση των ανθρώπινων ζώων είναι φυσικά η βασική προτεραιότητα. Ενώ λοιπόν θέλουμε πιο αποτελεσματική επιβολή του νόμου κατά των διακινητών και των λαθρεμπόρων, θα πρέπει να βρούμε ασφαλείς εναλλακτικές λύσεις σε αυτά τα επικίνδυνα ταξίδια και νόμιμες διάβλους, όπως την επανεκατάσταση, την ε, οικογενειακή επανένωση και την παροχή θεωρήσεων. Μάλιστα, ε, συναντήθηκα με ανθρώπους από τη Συρία, τη Βιανμάρ, το Αφγανιστάν και από το Κονγκό που ε, είχαν ε, επανεγκατασταθεί. Βέβαια και η νέα του ζωή είναι αρκετά δύσκολη, αλλά τουλάχιστον ε, ζουν με ασφάλεια. Και στο νέο τους σπίτι βρίσκουν βοήθεια και συμπαράσταση. Και έχω πολλά τέτοια παραδείγματα στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε πολύ περισσότερο όμως αυτούς τους καιρούς ιδιαίτερος. Σήμερα το πρωί είχα και μια άλλη ευκαιρία. Συνάντησα ένα κορίτσι από τη Συρία που είχε ξεφύγει από τις φρικαλαιότητες και τη βαναυσότητα στην πατρίδα της. Συγκινήθηκα τόσο πολύ όταν μου απέφθινε έκκληση αυτό το κορίτσι και μου παρουσίασε μου εξιστόρισε το όνειρό της και εγώ την ενθάρρυνα. Της είπα μην απελπίζεσαι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη είναι στο πλευρό της, στο πλευρό το δικό της και της οικογένειάς της και ολόκληρου του λαού της Συρίας. Η συνάντηση αυτή ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές για μένα. Αξιότιμη Ευρωβουλευτέ, Τα Ηνωμένα Έθνη χαιρετίζουν τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια σωστή κατάλληλη μεταναστευτική πολιτική. Και η σημερινή αναγγελία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πρόταση επανεκατάστασης 40.000 τον άσυλο είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Σας ενθαρρύνω λοιπόν σας τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπόνια στην εξέταση αυτής της σημαντικής πρότασης και να επιμεριστούν τις ευθύνες τους γιατί ένας επιτυχής επιμερισμός των ευθυνών θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένας επιτυχής επιμερισμός των ευθυνών θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει τη δραματική αύξηση των μεταναστευτικών ροών δίνοντα ταυτόχρονα ένα παράδειγμα προ μίμηση και για τι άλλε περιοχέ του κόσμου που αντιμετωπίζουν παρόμοιε προκλήσει. Τα Ηνωμένα Έθνη και η ΥΠΑΤΗ Αρμοστία για του πρόσφυγες, καθώ και διεθνεί οργανώσει ε, για τη μετανάστευση, θα συνεχίσουν τη συνεργασία του με τους Ευρωπαίους ηγέτες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κρίση με τρόπο ώστε ε, να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο. Η προσέγγιση μας θα πρέπει να είναι σφαιρική. Θα πρέπει να εξετάζουμε την κατάσταση και στις χώρες προέλευσης, διαμετακόμισης, διέλευσης και προορισμού. Και κυρίως θα πρέπει να διορθώσουμε τα αναπτυξιακά σφάλματα και τις συγκρούσεις που είναι οι αιτίε της μετανάστευσης. Πολύ περισσότερο από ό,τι τα τελευταία χρόνια και σχεδόν τόσο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επίσης θα πρέπει να αποφύγουμε τη, ε, τη στιγματοποίηση και τις διακριτικές, ε, τη διακριτική μεταχείριση εις βάρος των μεταναστών. Ταυτόχρονα έχουμε μία γύραση του πληθυσμού και ένα δημογραφικό πρόβλημα. Οπότε για να αντιμετωπίσουμε το έλλειμμα στο εργατικό δυναμικό μας και να διασφαλίσουμε τον οικονομικό μας δυναμισμό, στην, στην Ευρώπη χρειαζόμαστε τους μετανάστες. Η μεταπολεμική ιστορία της Ευρώπης δίνει ένα από τα πιο ιστορικά και θετικά παραδείγματα της συνεργασίας υπέρ της ειρήνης και της ευημερίας. Η ευρωπαϊκή επιτυχία έγινε πόλος έλξης για τους μετανάστες. Οι αξίες και οι κατευθυντήριες γραμμές και αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντικές. Γι' αυτό σας ενθαρρύνω να ανταπεξέλθετε το ύψο των περιστάσεων και τι υψηλέ προδιαγραφές που θέσατε για σας και για τον κόσμο ολόκληρο. Και θα έρθω τώρα στην ε, τρίτη σημαντική παγκόσμια πρόκληση για την οποία περιμένουμε τον ηγετικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε μια κρίσιμη χρονιά για την βιώσιμη ανάπτυξη. Πρέπει λοιπόν ε, να ε, χαρακτηριστεί αυτή η χρονιά από σημαντικές παγκόσμιες δράσεις. Και το 2015 θα έχουμε τρεις ιστορικές ευκαιρίες για να βάλουμε τον κόσμο σε ένα βιώσιμο, ε, ευήμερο και δίκαιο μονοπάτι. Η πρώτη ιστορική ευκαιρία θα είναι την 1η Ιουλίου, που θα πρέπει να ανανεώσουμε την παγκόσμια εταιρική σχέση για την ανάπτυξη στη διεθνή διάσκεψη ε, της χρηματοδότησης της ανάπτυξης που θα γίνει στην Αντίσα Μπέμπα. Οι ανεπτυγμένες χώρες ε, έχουν ευθύνη να πρωτοστατήσουν και να παράσχουν τα κονδύλια για την εξάλληψη της ακραίας φτώχειας και της εξαθλίωσης και την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, η ODA όπως τη λέμε, θα αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα και σημαντικό της ε, χρηματοδότησης κυρίως των λιγότερο ανεπτυγμένων χώρων και των μικρών νησιωτικών αναπτυσσομένων χωρών που χρειάζονται κατεπηγόντως συνεχή και μάλιστα και αυξημένη υποστήριξη και αρρωγή. Και οι χώρες που υλοποίησαν το στόχο της ε, αφιέρωσης του 0,7 του ΑΕΠ τους ε, στην επίσημη αναπτυξιακή ε, βοήθεια να το συνεχίσουν και 0,2% για τις, λιγότερες λιγότερο αναπτυγμένες χώρες είναι αυτός ο στόχος. Θα ήθελα να ενθαρρύνω όλες τις χώρες του ΩΣΑ να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα προς μίμηση. Και χθε ε, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανανέωσαν την απόφαση τους ε, και τη δέσμευσή τους υπέρ αυτού του στόχου. Ενθαρρύνω την Ευρωπαϊκή Ένωση να υλοποιήσει αυτό το στόχο το συντομότερο δυνατό. Επίσης, γνωρίζουμε ότι από μόνη της η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια δεν αρκεί. Θα πρέπει να βρούμε κονδύλια από πολλές πηγές και δημόσιες και ιδιωτικές. Η πρωταρχική ευθύνη της χρηματοδότησης της αηφόρου ανάπτυξης βέβαια έγκυται στις κυβερνήσεις. Γι' αυτό και θα πρέπει να στηρίξουμε την βελτίωση των δίκαιων εθνικών φορολογικών συστημάτων. Επίσης θα πρέπει να έχουμε ένα πιο έντονο παγκόσμιο μια πιο έντονη παγκόσμια φορολογική συνεργασία για να πατάξουμε τις παράνομες ε, διακινήσεις κεφαλαίων και την φοροδιαφυγή. Η διάσκεψη της Αντισαμπέμπα θα είναι κρίσιμη για τη δημιουργία εμπιστοσύνης, τη δημιουργία όθησης και, να, και την συμβολή της στην υλοποίηση των μελλοντικών μας στόχων. Το δεύτερο ορόσημο ε, θα έρθει το Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη. Εκεί οι χώρες ε, θα πρέπει να υιοθετήσουν ε, μια σημαντική, ένα σημαντικό θεματολόγιο για μετά το 2015 για τους νέους βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους, τα SDGs. Πρόκειται για ένα θεματολόγιο που θα έχει οικουμενικό χαρακτήρα και θα είναι φιλικό στους, προς τους πολίτες και στο περιβάλλον. Θα πρέπει να σταματήσει η μη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση στον κόσμο. Και εκεί θα μπορούσε να προταστατήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνουμε τη μετάβαση προς μια οικονομία που θα χρησιμοποιεί λιγότερο ε, άνθρακα. Επίσης, το Δεκέμβριο στο Παρίσι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ανανεώσουν την ε, δέσμευσή τους και να υιοθετήσουν μια οικουμενική συμφωνία υπέρ του κλίματος στην ε, συμφωνία, στη διάσκεψη για το περιβάλλον που θα λάβει η χώρα στο Παρίσι. Και εκεί η ηγετική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντική. Θα πρέπει να πρωτοστατήσετε στη λήψη μιας απόφασης για να αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές αλλαγές, να βελτιώσουμε την ευημερία, να ενισχύσουμε την ασφάλεια συμπεριλαμβανομένης και της ενεργειακής ασφάλειας. Και με τις εθνικές δεσμεύσεις αλλά και με την πολιτική της, την ενεργειακή, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προλιάνει το έδαφος ε, για να καταλήξουμε σε ένα ασφαλές ε, μέλλον πιο ευήμερο και με λιγότερη χρήση άθρακα. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί είναι ε, από τους πρώτους που το Μάρτιο ενίσχυσε αυτούς τους κλιματικούς στόχους και επίσης ε, είναι σημαντική και γενναιόδορη η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πράσινο Ταμείο για το Περιβάλλον. Η χρηματοδότηση είναι κέρια για να εξασφαλίσουμε μια φιλόδοξη συμφωνία στο Παρίσι. Θα πρέπει αυτή να είναι και πολιτικά αξιόπιστη για να μπορέσουμε να βρούμε τα 100 δισεκατομμύρια ετησίως που θέλουμε μέχρι το 2020 και το πράσινο το Ταμείο για το Κλίμα θα πρέπει να λειτουργήσει και πριν το Παρίσι για να βοηθήσει νησιωτικές ε, αναπτυσσόμενες χώρες, λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και τις αφρικανικές χώρες. Γι' αυτό και ζητούμε την ε, ισχυρή υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να εξασφαλίσουμε αυτό το στόχο. Επίσης, θα ήθελα να ζητήσω την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός ειδικού πακέτου για τις πλέον ευάλωτες χώρες, καθώς και τις νησιωτικές αναπτυσσόμενες χώρες και λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες τους ε, και από την άποψη του, των κλιματικών αλλαγών και από την άποψη της ανάπτυξης. Το πακέτο αυτό θα πρέπει να αφορά κυρίως τη χρηματοδότηση, την ανθεκτικότητα, την προσαρμογή και την ενέργεια. Και τέλος, θα ήθελα να παροτρύνω την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να πρωτοστατεί στις φιλόδοξες προσπάθειές της προκειμένου να ευοδοθεί μια φιλόδοξη συμφωνία στο Παρίσι και να ενισχυθούν οι κλιματικοί στόχοι για το 2020 και ταυτόχρονα να υιοθετηθούν πιο φιλόδοξοι στόχοι για την περίοδο μετά το 2020. Thank you for your support. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας, κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι βουλευτές. Είναι η 70η επέτειος φέτος των Ηνωμένων Εθνών. Η οργάνωσή μας γεννήθηκε από τις τάχτες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου που κατέστρεψαν μεγάλα τμήματα της Ευρώπης για την ειρήνη και την ευημερία, για ένα συγκεκριμένο σύμβολο των όσων πετύχαμε ακόμα και μετά τη μεγαλύτερη καταστροφή. Ζούμε σε ένα περίπλοκο κόσμο με πολλές προκλήσεις, αλλά πιστεύω ότι ζούμε και σε ένα κόσμο ευκαιριών και πιστεύω ότι είστε θεματοφύλακας λοιπόν των ευκαιριών αυτών. Ένας, μια ε, μηχανή και σας ε, καλώ να οθήσετε τον κόσμο με την κινητήριο αυτή δύναμή σας. Από κοινού μπορούμε να πετύχουμε έναν πιο δίκαιο κόσμο για την σημερινή και για την μεραντική γενιά και τις μελλοντικές γενιές. Σας ευχαριστώ για την δέσμευσή σας, για τη δημοκρατία και για το πνεύμα ευγένειας ε, και την εξυπηρέτηση των Ευρωπαίων πολιτών. Σας ε, ευχαριστώ για την υποστήριξη των ιδεών και των αξιών των Ηνωμένων Εθνών και για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας απευθύνω το λόγο. Εξοχότητες σας, ε, αξιότιμοι βουλευτές. Θα ήθελα από κοινού να διανύσουμε την απόσταση αυτή προκειμένου να γίνει ένας καλύτερος τόπος αυτός ο κόσμος όπου όλοι οι λαοί ανεξάρτητα από το που είναι μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια, όπου κανείς δεν θα μείνει πίσω. Αυτό είναι η πολιτική και ηθική επιταγή και ευθύνη. Η δική μου, η δική σας, η δική μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ηγεσία και την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γενική Γραμματέα. Καταλαβαίνετε γερμανικά, δεν χρειάζεστε διερμηνία. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ κύριε Γενική Γραμματέα. Νομίζω ότι η αντίδραση του Κοινοβουλίου σας έδειξε ότι τα θέματα τα οποία θίξατε είναι τα θέματα που μας απασχολούν και εμάς. Σας είμαστε ευγνώμονες για την δεύτερη αυτή επίσκεψή σας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και θα ήθελα να δράξω τη συγκεκριμένη ευκαιρία, λοιπόν, κύριε Γενική Γραμματέα, για να σας αναφέρω ότι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, νομίζω ότι μπορώ να το πω εξ όλων των συναδέλφων, όχι μόνο ευχαριστούν τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά και εσάς προσωπικά γιατί πιστεύω ότι είσαστε ένας από τους αξιόπιστους εκπροσώπους της ιδέας της ειρηνικής συνεργασίας των λαών στον πλανήτη. Γι' αυτό λοιπόν και προσωπικά σας απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ κύριε Γενική Γραμματέα.